Right, good afternoon, ladies and gentlemen. It's 12 minutes past three. We're running late. We better start. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινήσουμε γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο. Υπαριθμόν 1, σημείο στη μερίσια διάταξη, έγκριση, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις την εγκρίνουμε. Σημείο 2, ανακοινώσει του Προέδρου. Να σας κάνω κάποιες σύντομες ανακοινώσεις. Στις 8 Οκτωβρίου, οι συντονιστές της Επιτροπής μας ενέκριναν την αξιολόγηση που θα πρέπει να υποβληθεί στον Πρόεδρο μετά την ακρόαση του κυρίου Μπορέλ, που, είναι υποψήφιος για τη θέση του ΥΠΑ του εκπροσώπου για τις εξωτερικές υποθέσεις και τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε λάβει περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τις εκκρεμούσες υποψηφιότητες. Ο κύριος Σασόλη μας είπε σήμερα ότι η έγκριση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενδεχομένως να παραταθεί μέχρι την 1η Δεκεμβρίου βάσει του χρόνου που απαιτείται προκειμένου οι απομείνασε χώρε να υποβάλουν υποψηφιότητε. Αυτή τη στιγμή οι τρει αυτοί υποψήφοι υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα γίνει μια σειρά νέων αξιολογήσεων και τότε θα είμαστε σε θέση να γνωρίσουμε ακριβώ και πότε θα γίνουν αυτέ οι αξιολογήσει. Σήμερα, την Τετάρτη αυτή στι 3 το μεσημέρι, θα συνεδριάσει διάσκεψη των Προέδρων, η οποία θα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό περαιτέρω. Ζήτησα από τη Γραμματεία πάντω να σα κρατήσει ενήμερου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν νέε εξελίξει για το ζήτημα αυτό του διορισμού τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημείο 3 τη ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσει του Προέδρου σχετικά με τι αποφάσει που έλαβαν συντονιστέ βάσει του κανόνα 214 του κανονισμού μας στις 13 ε, Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα των συντονιστών. Έχετε στην ιστοσελίδα της ΑΦΕΤ ε, τα πρακτικά και τα συμπεράσματα της συνεδρίασης αυτής και θα συμπεριληφθούν επίση και στα πρακτικά τη σημερινή η Σημείο 4 τη ημερήσια διάταξη. Τα σημεία 4, 5, 6 και 7 μπορούν να συζητηθούν από κοινού, γιατί όλα έχουν να κάνουν με τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή μα όσον αφορά τη σύναψη μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και μια συμφωνία προστασία των επενδύσεων μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Βιετνάμ. Τι γνωμοδοτήσει αυτέ τι ζήτησε η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η σύνταξη της γνωμοδότησης αυτή θα γίνει βέβαια σε στενή συνεργασία με τη δική μας την Επιτροπή. Η κυρία Λίμα που είναι η συγγήτρια συμμετέχει και στις δύο επιτροπές. Αυτό είναι θετικό. Θα μας παρουσιάσει ένα σύντομο κείμενο το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση των, του σχεδίου γνωμοδότησης όσον αφορά την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και τη Συμφωνία Προστασίας των Επενδύσεων μεταξύ τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βιετνάμ. Ιζαμπέλα, μάλλον Προτού σας δώσω το λόγο, έχουμε ένα διαδικαστικό. Ένα λεπτάκι, σας το συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να θέσω ένα διαδικαστικό θέμα. Έχουμε την πρώτη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τη στιγμή αυτή που μιλάμε, μια όμορη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωση, η Τουρκία, στην οποία δίνουμε δισεκατομμύρια ευρώ, εισβάλλει σε μια όμορη τη χώρα, μια γειτονική της χώρα, τη Συρία. Υπάρχουν ε, χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες οι οποίοι εισβάλλουν αυτή τη στιγμή στη Συρία και προχωρούν σε ε, αιματοχυσίες άμεσες επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε εμείς να επιληφθούμε του ζητήματος αυτού και να μην συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τον συνήθι τρόπο business as usual. Σαφώς οφείλουμε να επιληφθούμε του ζητήματος αυτού καθότι είμαστε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πραγματικά οι ε, Ευρωπαίοι πολίτες δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν αυτή τη στιγμή αν δεν ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό που είναι ένα καυτό ζήτημα της επικαιρότητα. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που κάνει την εισβολή αυτή στη Συρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει να επιληφθεί του ζητήματος και να αποφανθεί επ' αυτού η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Καταρχάς δεν είμαστε σε business as usual κατάσταση. Έχω έρθει σε επαφή με το επιτελείο της κυρίας Μογκερίνη. Εκείνη, ενώ σήμερα είμαστε εμεί εδώ, βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, στο, στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών και ζήτησε από το επιτελείο τη, μόλι προκύψει κάποιο αποτέλεσμα από τη Σύνοδο αυτή των Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο, να ε, ενημερωθώ σχετικά με το περιεχόμενο να σας ενημερώσω βεβαίως και σας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αν γίνει κάτι τέτοιο. Είχαμε βεβαίως και την ιδέα να προσκαλέσουμε κάποιον από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για το ζήτημα αυτό σήμερα. Ωστόσο, επειδή γίνεται αυτή η σύνοδος στο Λουξεμβούργο, ε, δεν θα ήταν ε, ο καταλληλότερος τρόπος. Το σημειώσαμε, βεβαίως όλους μας απασχολεί. Βλέπω και ότι οι συνάδελφοι ε, συγκεντρώνουν υπογραφές. Πολλές πολιτικές ομάδες έχουν ήδη τοποθετηθεί επί του ζητήματος. Θα έλεγα το εξή. μόλις ενημερωθούμε από την ύπατη εκπρόσωπο, θα σας ενημερώσω εσάς και βεβαίω θα, θα θέσουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη κάποιας επόμενης συνεδρίας ή της επόμενης επόμενης συνεδρίασης. Απλά η τη επομενη συνεδριασης απλα η σημερινη μας συνεδρίαση γίνεται ταυτόχρονα με αυτή τη σύνοδο στο, στο Λουξεμβούργο. Γι' αυτό και δεν το θέσαμε το θέμα. Συνεχίζεται η σύνοδο αυτή γιατί ε, ξέρω ότι και ο Ουκρανός προσκεκλημένος μας είναι ακόμη στο Λουξεμβούργο. Ε, ίσως θα μπορούσαμε από εκείνον να ε, πάρουμε κάποιες πρώτες πληροφορίε ή από τον Υπουργό Εξωτερικών τη Βόρεια Μακεδονίας που θα έχουμε σήμερα μαζί μας. Ε, σε κάθε περίπτωση το καταγράφουμε βεβαίω και δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε. Και άλλο διαδικαστικό θέμα. Παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο μιλητής. Σημείο 3. Αναφέρομαι στο σημείο 3. Στη διάρκεια της συνεδρίασης των συντονιστών ε, δόθηκαν 13 ε, εκθέσεις για την γειτονία και για την ενταξιακή διαδικασία. Αυτές οι 13 εκθέσεις κατανεμήθηκαν ανάμεσα σε τρεις μονάχα ομάδες, δηλαδή ούτε η CR ούτε η GUE, ε, ούτε το IDE πήραν καρμία έκθεση. Έστειλα επιστολή προς τον Πρόεδρο και ρώτησα γιατί. Διακόπτει ο πρόεδρο. Κύριε Μαγιανή, ήδη μου στείλατε το mail. Ναι, μάλιστα, και το διάβασα ήδη λέει ο πρόεδρος, και έχω δει τουλάχιστον ένα σχέδιο απάντησης. Το, άρχισα να το ετοιμάζω το Σαββατοκύριακο. Το στείλατε ήδη? Σας έχω στείλει ήδη απάντηση. Μάλ. Ναι, γαλλογερμανική αποτελεσματικότητα. Ναι, αλλά Ελπίζω πως μετά θα αυτό θα είναι και η γαλλική ισότης για όλες τις ομάδες. Εγώ σας έχω αναφέρει όλα τα επιχειρήματα. Οι αποφάσεις αυτές ελευθύσαν από τις πολιτικές ομάδες. Έχουμε τον κανόνα αυτό ότι οι ομάδες μπορούν να αποφασίζουν μεταξύ τους. Κατανοώ ποια είναι η ανησυχία σας. Ίσως να θυμάστε ότι έκανα και ένα σχετικό σχόλιο στην Επιτροπή των Συντονιστών. Θα τα πάρετε όλα γραπτό. Ίσως μπορείτε τώρα να ελέγξετε τα mail σας. Εντάξει, μπορώ να περιμένω άλλη μια μέρα. Και συνάδελφε Μαριανή, ε, προτείνω στην επόμενη σύνοδο των συντονιστών να ε, ασχοληθούμε και πάλι με αυτό το θέμα. Άλλα θέματα διαδικαστικά, όχι, οπότε ερχόμαστε τώρα στο σημείο 4 και θα δώσω το λόγο στην κυρία Ιζαμπέλ Βίσλερ Λίμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω θα ε, να πω ότι όντως σήμερα δεν μπορούμε να παρεστάνουμε ότι δεν τρέχει τίποτα γιατί στο μυαλό μας όλοι έχουμε αυτό που συμβαίνουν στη Συρία. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω αυτήν το σχέδιο γνωμοδότησης της ΑΦΕΤ για την σύναψη της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ και ε, της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ. Υπάρχει σαφώς δεσμός ανάμεσα στην, ε, στην, στην, Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας και της, Ευρωπα... και της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών, όπου τα δύο μέρη ε, υπόσχονται να τηρούν τις ε, υποχρεώσεις τους ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ε, εφαλτήριο για και έναν γνώμονα για παρόμοιες συμφωνίες αναπτυσσόμενων χωρών, αναδυόμενων χωρών της περιοχής. Το Βιετνάμ είναι ένα κατεξοχήν εταίρο στην Νοτιοανατολική Ασία, ιδιαίτερα όσον αφορά τι διαπραγματεύσει για τι κλιματικέ αλλαγέ, τη χρηστή διαχείριση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, καθώ και την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Το Βιετνάμ έχει καταβάλει προσπάθειε για να κάνει σημαντικέ και φιλόδοξε μεταρρυθμίσει, ιδιαίτερα όσον αφορά το περιβαλλοντικό δίκαιο και το εργασιακό Εργασιακό Δίκαιο καθώς και έχει κυρώσει έξι από τις οχτώ ε, βασικές συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Ωστόσο, παραμένει ανησυχητική η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά η εφαρμογή της ε, θανατικής ποινής. Πρέπει το Βιετνάμ να προχωρήσει προς ε, μορατόριο και κατάργηση. η αξιολόγηση του αντικτύπου αυτής της συμφωνίας θα πρέπει να γίνεται περιοδικός. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο άρθρο 13 της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών, όπου ε, μιλάμε για συνεργασία επί τη βάση κοινών αξιών και αρχών, λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα ανάπτυξης των δύο μερών. Θα πρέπει να υπάρχει κατά τη γνώμη μου ένας μηχανισμός που θα αντιμετωπίζει θέματα διαφορών. Και γι' αυτό καλωσορίζω ότι η πιθανότητα επίλυση διαφορών υπό το άρθρο 13 για την ε, εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη και από την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης σε περίπτωση που δεν λυθούν τα, οι διαφορές υπάρχει και δυνατότητα ενός δεύτερου μηχανισμού που επιτρέπει στο ένα μέρος να ε, ζητήσει τη σύσταση ενός ανεξαρτήτου πάνελ υπερηγνωμόνων για να εξετάσει το θέμα. Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ πως η συμφωνία μας παρέχει τη δυνατότητα μόχλευσης που μπορεί να αξιολογήσει την πρόοδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είμαστε ανοιχτοί και θέλουμε να διατηρήσουμε ε, ε, τη δυνατότητα να θίξουμε το, τα, τα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά την Συμφωνία Επενδύσεων, να πούμε ότι αυτά τα εργαλεία είναι σημαντικά για τη βελτίωση της διαβίωσης των λαών. Ένας από τους στόχους αυτής της συμφωνίας είναι να ενισχυθούν οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ένωσης και Βιετνάμ, σύμφωνα με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και να προωθήσει το εμπόριο και τις επενδύσεις υπ' αυτή την συμφωνία λαμβάνοντας υπόψη βέβαια τα περιβαλλοντικά στάνταρ και τις διεθνείς συμφωνίες. Όσον αφορά την προστασία δε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήθελα να τονίσω ότι το άρθρο 35 της Συμφωνίας Εταιρική Σχέσης και Συνεργασίας ανάμεσα στην Ένωση και το Βιετνάμα. σύμφωνα με αυτό το άρθρο, τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των οποίων είναι συνυπογράφοντα μέρη. Η συμφωνία για τις επενδύσεις έχει τη δυνατότητα να, να βελτιώσει τα συνθήκες διαβίωσης, να προωθήσει την οικονομία, τη χρηστή διαχείριση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το Βιετνάμ και να προωθήσει τους στόχους ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Γι' αυτό και πιστεύω πως θα πρέπει να εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη δε το περιορισμένο αριθμό ε, σελίδων για αυτή τη γνωμοδότηση θα προσθέσω κάποιες τροπολογίες και θα ήθελα να ευχαριστήσω δε το επιτελείο του, ε, του ΕΛΚ και τους βοηθούς μου για την ε, βοήθεια που μου προσέφεραν σύνταξη αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ, πολύ κυρία Λίμα. Έχουμε κάποια λεπτά πριν να φτάσει ο Υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας. Ποιος θέλει πρώτος το λόγο? Ο κύριος Κοτσολίνο. Πού είστε? Α, εκεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μιλώ εξ ονόματος του κυρίου Βούτσμαν που είναι σκιώδης σε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση. Όπως ήδη υπογραμμίστηκε θα υποβάλλουμε διάφορες τροπολογίες για να τονίσουμε τις πολυάριθμες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και την ανεπάρκεια των εγγυήσεων ε, σχετικά με αυτό το θέμα. Ας πούμε εκφοβισμοί, κρατήσεις, υψηλό αριθμό εκτελέσεων ε, των συνδικαλιστών ηγετών, των ακτιβιστών, ακόμα και μετά την έναρξη της συμφωνίας ισχύου αυτής της ε, συμφωνίας. Για το κεφάλαιο ε, δε ε, βιώσιμης ανάπτυξης δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πρόοδο λόγω του δεν υπάρχει οδικός χάρτης θα πρέπει να ζητήσουμε τη δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού παρακολούθηση για να αξιολογούμε διαρκώς την κατάσταση στη χώρα, να ζητάμε την απελευθέρωση των, πολιτικών κρατούμενων, την ανεξάρτητη εκτίμηση της των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και ε, την ύπαρξη των απαραίτητων συνθήκων για να δώσουμε την έγκρισή μας προς αυτή την έκθεση. Επίσης, η έλλειψη έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα μας οδηγεί στο να ζητήσουμε από την Κομισιόν μια αξιολόγηση της κατάστασης πριν να δώσουμε την έγκρισή μας για την συμφωνία αυτή. Θα υποβάλουμε λοιπόν οι σοσιαλιστές τροπολογίες και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπο πλήρους συνεργασίας με την εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Speakers, Mr. Ράιουσεν. Ο κύριος Ράιουσεν, εκ μέρους του ECR. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βίζελε Λίμα για το σχέδιο της γνωμοδότησης. νομίζω ότι θέτει τον δάκτυλο επί το τύπο των ήλων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ προβληματική. Το Βιετνάμ είναι μια χώρα όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ε, ε, παντοδύναμο. Από το 1953 δεν έχουν γίνει ελεύθερες εκλεγές, δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης, δεν υπάρχει ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης. Ασκούνται τεράστιες πιέσεις σε αυτές τις ε, ελευθερίες. Οι χριστιανοί θεωρούνται ως πράκτορες των ξένων ε, θεωρούνται απειλή για τη χώρα και αποκλείονται από την συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική ζωή. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα στο Βιετνάμ το 2019. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα σε αυτό το μέτωπο και πρέπει να αναλάβει πολύ ισχυρότερε δράσει εναντίον του Βιετνάμ σε αυτά τα ζητήματα. Η Συμφωνία ε, Ελευθέρων Συναλλαγών ξεκινά έναν διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καλό είναι αυτό. Φυσικά Καλό είναι το ότι υπάρχει μια τέτοια πρόβλεψη. Αλλά το ερώτημα είναι, επαρκεί μια τέτοια πρόβλεψη από μόνη τη. Ενδεχομένως να μην αρκεί να μιλάμε απλώς, να κάνουμε διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ίσως αυτές τις εμπορικές συμφωνίες θα έπρεπε να προσπαθούμε να εντάσσουμε πιο δεσμευτικά μέτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε εδώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ο κύριος ε, Μιχαήλ Γκάλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Μιλάμε προφανώς για μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών και για μια συμφωνία προστασία ε, των επενδύσεων που βεβαίως πηγαίνουν χέρι-χέρι πάντοτε. Λογικό είναι. Τίθεται λοιπόν το θεμελιώδες ερώτημα αν αυτή η συμφωνία πρόκειται να οδηγήσει στον δημοκρατικό μετασχηματισμό της χώρας. Ε, η απάντηση είναι προφανώς όχι. Με μια εμπορική συμφωνία δεν μπορεί κανείς να θέσει τέλος στην παντοδυναμία ε, του Κομμουνιστικού Κόμματος, ούτε να ε, δημιουργήσει μια δημοκρατία, ένα επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έτσι όπως θα το επιθυμούσαμε εμείς. Όμως δεν είναι αυτό το, το αποφασιστικό σημείο. Διότι το ερώτημα που επίση τίθεται είναι αν δεν γίνει μια τέτοια συμφωνία θα αυξηθούν οι δυνατότητε μα ε, όσον αφορά την, να ασκήσουμε επιρροή σε αυτή τη χώρα. Επίση όχι. Γιατί νομίζω ότι με αυτή τη συμφωνία ε, αποκτούμε, χτίζουμε γέφυρε με τη χώρα αυτή, μέσα από τι οποίε θα μπορέσουμε να επιδιώξουμε ακριβώ αυτά που επιθυμούμε στον τομέα των ε, εργασιακών δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη προστασία του περιβάλλοντο. Τότε εξασφαλίζουμε αυτή τη δυνατότητα, αν συνάψουμε τη συμφωνία αυτό. Φυσικά, ξαναλέω, η κατάσταση δεν πρόκειται να, μας, να, ε, να, είναι ιδανική, δεν πρόκειται να, να οδηγηθούμε σε μια ιδανική κατάσταση. Όμως το, το, το γεγονός ότι 6 από τις 8 βασικές συμβάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας έχουν πλέον επικυρωθεί, ε, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, ένα βάθρο αν θέλετε, για να προχωρήσουμε τον διάλογο σε αυτά τα ζητήματα τα εργασιακά και στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, ε, ε, προβλέπονται και πολύ φιλόδοξες μεταρρυθμίσει όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, ε, που επίσης εντάσσονται και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτής της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών. Στην γενική στάθμιση λοιπόν του ερωτήματος, ε, αν θα πρέπει να συνάψουμε μια τέτοια ε, συμφωνία ή όχι, εγώ δηλώνω ξεκάθαρα ότι είναι καλύτερα να συνάψουμε μια τέτοια συμφωνία και γι' αυτό σας καλώ συνάδελφοι να υποστηρίξουμε αυτή την προοπτική. Ευχαριστώ. Η κυρία Λαζό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο κύριο Γκάλερ. Όλοι γνωρίζουμε πώ έχει η πολιτική κατάσταση στο Βιετνάμ. Δεν πρόκειται για μια νέα πολιτική κατάσταση. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει είναι η δική μας ικανότητα ως Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσουμε περισσότερο και με έναν τρόπο πιο ηχηρό τις αξίες μας. Είτε πρόκειται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε πρόκειται για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να αδιαφορήσουμε μπροστά στην υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας με το Βιετνάμ, γιατί στην περίπτωση αυτή αφήνουμε ένα κενό και ουσιαστικά προωθούμε ή σπρώχνουμε το Βιετνάμ να επιλέξει άλλους εταίρους. Το σημαντικό είναι λοιπόν να υπογράψουμε τις δύο αυτές συμφωνίες, αλλά εφαρμόσουμε αυστηρά τις δύο αυτές συμφωνίες με όλες τις ρήτρε, ακόμα και με τις ρήτρε αναστολής που προβλέπονται, αν τυχόν προκύψουν σημαντικά προβλήματα. Επ' αυτού έχω εγώ ακόμα κάποιες ανησυχίες και κάποιους ενδιασμούς ως προς το πώς έχουν συνταχθεί οι δύο αυτές συμφωνίες. Σαφώς το περιεχόμενο είναι σωστό, αλλά θα πρέπει να μπορεί να επιτρέπει και οι συμφωνίε αυτέ να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε προφανώς να μπορούμε μέσω του εμπορίου να εξάγουμε και τις αρχές μας και τις θεμελιώδεις αξίες μας προς το Βιετνάμ. Σίγουρα το χειρότερο σενάριο θα ήταν να μην υπογράψουμε τις συμφωνίες αυτές και να αφήσουμε τελικά το Βιετνάμ να επιλέξει να υπογράψει εταιρικέ σχέσεις με άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν τους ίδιους στόχους με εμάς όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ή την βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστούμε για την ομάδα ID ο κύριος Ριβιέρα. Ριβιέρ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Βιετνάμ γνωρίζετε ότι είναι μια πολύ σημαντική πλατφόρμα εξαγωγής κινέζικων προϊόντων. Το να συνάψουμε λοιπόν αυτές τις δύο συμφωνίες με το Βιετνάμ ουσιαστικά ε, συνεπάγεται με μία λευκή επιταγή προς την Κίνα να εξάγει χωρίς κανένα εμπόδιο, χωρίς κανένα περιορισμό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από αυτό θα ήθελα να επανέλθω σε ένα σημείο που θίξανε και οι προλαλήσαντες. Το ότι υπολείπεται πάρα πολύ το Βιετνάμ όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όλος ιδιαιτέρως θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των μελών της Επιτροπής μας στην ε, ελευθερία θρησκευτικών πεπιθήσεων. Οι χριστιανοί είναι αυτοί οι οποίοι επί του παρόντος είναι θύματα καταστολής στην δημοκρατία του Βιετνάμ. Βλέπουμε όλο και περισσότερο τέτοιες καταστάσεις και σε άλλες χώρες, πέρα από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Νομίζω δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την περίπτωση του κύριου Βαγγινελή, ο οποίος είναι μια προβεβλημένη προσωπικότητα της Καθολικής Εκκλησίας στο Βιετνάμ. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής να λάβουμε υπόψη μας και την πολιτική που ακολουθεί το Βιετνάμ όσον αφορά τα στι θρησκευτικέ πεπιθήσει, όπου δεν αναγνωρίζεται τελικά κανένα δικαίωμα ελευθερία πεπιθήσεων και ανεξιθρησκεία. Πρόεδρο. Σα ευχαριστούμε. Δεν νομίζω θέλει να πάρει κανεί άλλο το λόγο. Επομένω, Ιζαμπέλα, θέλετε να απαντήσετε. Ναι, θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που έχει υπογραφεί πλέον η συμφωνία και όπου εμείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα, τα περιορισμένα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προφανώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μοχλό που έχουμε στη διάθεσή μας για να σημειώσουμε πρόοδο, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι συμφωνίες αυτές έχουν υπογραφεί. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας, ουσιαστικά στέλνουμε σε ελληνικές καλένδες και τις δύο αυτές συμφωνίες. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ πάντω για τι παρεμβάσει σα και προσβλέπω σε μια επικοδομητική συνεργασία με όλου όσοι επιθυμούν να σημειώσουμε πρόοδο για τι δύο αυτέ γνωμοδοτήσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία και εμεί σα ευχαριστούμε. Με ενημέρωσαν ότι εκπρόσωπος από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εδώ, η κυρία Ντάλι και Μπέρτς συγκεκριμένα. Επιθυμείτε να πάρετε το λόγο εν συντομία. πρώτος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που μας προσκαλέσατε να συμμετάσχουμε στην σημερινή συζήτηση, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Βιετνάμ βελτιώνονται όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό το είδαμε και στο πλαίσιο της διαπραγμάτευση διαφόρων συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των δύο αυτών συμφωνιών που ε, εξετάζουμε στην Επιτροπή σας σήμερα. Πάντως ε, και αργότερα αυτή την εβδομάδα ελπίζουμε ότι ε, οι εκπρόσωποι μας θα υπογράψουν μία ακόμα συμφωνία με το Βιετνάμ που θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα αυτή να συμμετέχει περισσότερο σε κάποια προγράμματα ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένες αποστολές Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι βελτιώνονται σταθερά οι σχέσεις μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις διμερείς μας σχέσεις με το Βιετνάμ, αλλά και εν γέννη για όλη την περιφέρεια, καθότι το Βιετνάμ διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα πλαίσια του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Άζιαν και μάλιστα του χρόνου θα προεδρεύει της Άζιαν το Βιετνάμ. Βέβαια δεν κινήθηκαν τα πάντα ομαλά και εύκολα το τελευταίο διάστημα. Σαφώς αντιμετωπίσαμε δύσκολες καταστάσεις, εντάσεις μεταξύ αυτών που είναι πιο φιλελεύθεροι και διαλλακτικοί και αυτών οι οποίοι διατηρούν μια πιο σκληρή, σκληροπυρηνική στάση, τόσο στο πλαίσιο της κυβέρνησης και στο πλαίσιο του ίδιου του κόμματος. Πάντως υπάρχουν ε, όντως πολλά στοιχεία τα οποία μπορούν να επηρεάσουν ε, την ε, διαπραγμάτευση των συμφωνιών αυτών και θεωρούμε ότι οι συμφωνίες αυτές, σαν αυτές που εξετάζουμε τώρα, πραγματικά ενισχύουν όλους όσους θέλουν να έχουν ένα Βιετνάμ το οποίο θα είναι πιο διαλλακτικό και πιο ανοιχτό προς τον έξω κόσμο και νομίζω ότι μέσω των δύο αυτών συμφωνιών μας δίνεται πραγματικά η δυνατότητα ω Ευρωπαϊκή Ένωση να διαβιβάσουμε προς το Βιετνάμ περισσότερο τις δικές μας εισαρχέ, να καταφέρουμε να επηρεάσουμε θετικά κατά αυτόν τον τρόπο το Βιετνάμ. Προφανώς υπάρχουν αρκετά προβλήματα και ένα από αυτά, ένα πολύ σημαντικό είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα πολύ ευρύ τομέα. Υπάρχει ένας διάλογος επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το Βιετνάμ και μας δίνεται έτσι η δυνατότητα να θίξουμε συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την ίδια την κυβέρνηση των Βιετνάμ, η οποία αν δεν υπήρχε ο διάλογος αυτός δεν θα συζητούσε ποτέ τα ζητήματα αυτά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μα μα επιτρέπουν πραγματικά να δημιουργήσουμε καλύτερε συνθήκε μόχλευση υπέρ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντα και τα εργαλεία που έχουμε στα πλαίσια του ΠΟΕ και τα εργαλεία τα οποία προκύπτουν από την ίδια τη διαπραγμάτευση των δύο αυτών συμφωνιών, ελεύθερων συναλλαγών αλλά και τη Συμφωνία Προστασία των Επενδύσεων. Και θα χρησιμοποιήσουμε τη μόχλευση και τα εργαλεία αυτά και κατά την εφαρμογή των δύο αυτών συμφωνιών. Το Βιετνάμ εξελίχθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια, έχει καλύψει σημαντικό δρόμο και καθώς ανοίγει όλο και περισσότερο την οικονομία του προς τον έξω κόσμο, προφανώς προκύπτουν και ζητήματα τα οποία θα πρέπει εμείς να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγις. Όπως για παράδειγμα η στάση του Βιετνάμ απέναντι στη χρήση του διαδικτύου, απέναντι στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η στάση που διατηρεί η κυβέρνηση του Βιετνάμ όσον αφορά το ζήτημα της ελευθερίας της έκφρασης. Όλα αυτά, αν θέλετε, είναι νέα ζητήματα, πρωτόγνωρα ζητήματα για το Βιετνάμ. Έτσι λοιπόν μέσω όλων αυτών των συμφανιών αλλά και μέσω των διαφορετικών διαλόγων που έχουμε με το Βιετνάμ ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε να το πείσουμε να σέβεται περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα και να διορθώσει τα προβλήματα αυτά τα οποία έχουμε εντοπίσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας ακούσουμε τώρα και τον κύριο Μπέρτς από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο διάμεσο διάστημα μπορώ να καλωσορίσω επίσης και τον Υπουργό Δημητρόφα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα μιλήσω αγγλικά, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Θα είμαι σύντομο γιατί οι προλήσαντε κάλυψαν πολλά από τα ζητήματα που ήθελα να θίξω. Όντω, στα τέλη Ιουνίου υπεγράφησαν οι δύο αυτέ σημαντικέ συμφωνίε που το λένε πραγματικά ορόσημο στι σχέσει που έχουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση με το Βιετνάμ. Αν επικυρωθούν οι δύο αυτέ συμφωνίε, θα καταφέρουμε να έχουμε προτιμησιακή προσέγγιση σε μια οικονομία 100 εκατομμυρίων περίπου πολιτών, μια πολύ εύρωστη οικονομία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και στο πλαίσιο τη Άζιαν. Νομίζω λοιπόν ότι οι συμφωνίες αυτές θα μας δώσουν τη δυνατότητα να προωθήσουμε περισσότερο εμπορικές επενδύσεις, να αυξήσουμε τις εμπορικές συναλλαγές και να αυξήσουμε τις θέσεις απασχόλησης και στις δύο πλευρές, και στο Βιετνάμ δηλαδή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια το Βιετνάμ έχει γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός μας εταίρος μετά την Σιγκαπούρη στο πλαίσιο της Νοτιοανατολικής Ασίας και θεωρούμε ότι μέσω των συμφωνιών αυτών θα καταφέρουμε να καταρρύψουμε όλα τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν στο εμπόριο, θα ενισχυθούν οι διμερείς εμπορικές μας σχέσεις και οι εξαγωγές προς το Βιετνάμ θα αυξηθούν κατά 30%, ενώ οι εξαγωγές του Βιετνάμ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξηθούν κατά 20%. Και μακροπρόθεσμα όμως μπορούμε να έχουμε πολύ θετικέ εξελίξεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την γενικότερη δέσμευσή μα στην περιοχή της ASEAN και μετά την Σιγκαπούρη και την σχετική συμφωνία που έχουμε με τη χώρα αυτή, η συμφωνία που έχουμε αυτή τη στιγμή που θα έχουμε μάλλον με το Βιετνάμ θα είναι η δεύτερη πιο σημαντική συμφωνία που πραγματικά καταδεικνύει ότι δεσμευόμαστε όλο και περισσότερο με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Τα οικονομικά πλεονεκτήματα ουσιαστικά θα συνοδευτούν από νομικές δεσμεύσεις όσον αφορά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος προβλέπονται ως οριζόντιες αρχές οι ρήτρε αυτές και στο προήμιο των συμφωνιών αυτών, αλλά και στο συγκεκριμένο κεφάλαιο που έχει να κάνει με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Προβλέπονται συγκεκριμένε υποχρεώσει, δηλαδή όσον αφορά τα εργατικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από τι συμβάσει τη Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Και επίση προβλέπονται συγκεκριμένε περιβαλλοντικέ αλλά και κοινωνικέ υποχρεώσει που θα πρέπει να τηρήσει το Βιετνάμ, καθώ επίση και ε, η καταπολέμηση Τη κλιματικής αλλαγή. Προβλέπεται επίσης ένας μηχανισμός επίλυση των εμπορικών διαφορών και έχουμε δει ότι το Βιετνάμ ήδη προτίθεται να εφαρμόσει όλες τι απαραίτητε πολιτικές για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσει αυτές και έχει ήδη επικυρώσει μια σημαντική σύμβαση του διεθνού της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Πάντως αυτή τη στιγμή ε, η Εθνοσυνέλευση του Βιετνάμ προβλέπει μία τροποποίηση τη σχετική νομοθεσία που έχει να κάνει με το εργατικό δίκαιο, προκειμένου να συμμορφώνεται περισσότερο με τη Σύμβαση 98 τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία για τι Συλλογικέ Συμβάσει. Τώρα, όσον αφορά τις σχέσεις με την Κίνα. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών προβλέπονται πολύ αυστηροί και συγκεκριμένοι κανόνες όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής. Θα είναι απόλυτα σαφές δηλαδή για το τι αποτελεί προϊόν του Βιετνάμ, τι αποτελεί προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιο θα είναι το περιεχόμενο των προϊόντων αυτών και ποιο είναι το επίπεδο μεταποίησης το οποίο προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. Όλα αυτά ρυθμίζονται από τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και από ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο το οποίο έχει ως στόχο να αποφύγει οποιαδήποτε καταχρηστική μεταχείριση των πολιτικών που προβλέπονται για τους κανόνες καταγωγής. Θα έχουμε τη δυνατότητα στο σύντομο χρονικό διάστημα να συζητήσουμε περισσότερο με το Βιετνάμ, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της επικύρωσης των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Όπω σα είπα, έχουμε ήδη μια συμφωνία εταιρική σχέσης και συνεργασία. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται ότι η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και η Συμφωνία Προστασίας των Επενδύσεων θα έρθει να συμπληρώσει το πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε με το Βιετνάμ. Θα μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να έχουμε μια αμοιβαία εποφελή σχέση με το Βιετνάμ. Προφανώς το ζήτημα της εφαρμογής είναι πάρα πολύ σημαντικό και η ε, νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προβλέψει τη δημιουργία ενός νέου πεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα επιβλέπει πραγματικά την ορθή εφαρμογή των δύο αυτών ε, συμφωνιών. Όπως σας είπα, για τις δύο αυτές συμφωνίες θα θέλαμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα, ένα πλαίσιο επικοδομητικής συνεργασίας με το Βιετνάμ, προκειμένου να εμβαθύνουμε περισσότερο τη σχέση μας και σε κάθε περίπτωση η εναλλακτική, όπως υπόθηκε, θα ήταν να δημιουργήσουμε ένα κοινό και να προωθήσουμε τελικά, να σπρώξουμε το Βιετνάμ να συνεργαστεί με άλλες χώρες και όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να εγκριθούν αυτές οι δύο συμφωνίες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Νομίζω ότι ήταν ε, πολύ πολύτιμες οι πληροφορίες αυτές που ακούσαμε. Να σας ενημερώσω ότι το σχέδιο γνωμοδότησης θα ε, διαβιβαστεί στα μέλη των Επιτροπών ΑΦΕΤ και ΝΤΡΟΑ ε, το συντομότερο. Προθεσμία καταβολής τροπολογιών είναι η 11η Νοεμβρίου, 5 το απόγευμα και το σχέδιο γνωμοδότησης θα παρουσιαστεί 6 και 7 Νοεμβρίου στην ΑΦΕΤ. 8. Σημείο 8 της της διάταξης. Νικόλα, θέλεις να ανέβεις στο βήμα.